Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι καθίστε. Σας παρακαλώ καθίστε, λέει ο πρόεδρος Σούλτς. Προχωρούμε στην ψηφοφορία κυρίες και κύριοι. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ επί διαδικαστικού. Έχετε ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, έχει περάσει πάνω από μήνας από τότε που εδώ στο Κοινοβούλιο αποκαλύφθηκε η εκλογική απάτη, ή ε, μάλλον η απάντηση ως προς την ψηφοφορία της κυρίας Λεπέν. Ε, ε, διεξάγετε εσείς μια έρευνα. Θα θέλαμε να ξέρουμε, να γίνει ένας